Ελπίζω με αυτή την έκθεση του κυρίου Ντεζίρ να ακολουθήσει ένα νέο δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να γενικευθούν οι κανόνε, να γενικευθεί η εφαρμογή των κανόνων περί κοινωνική εταιρική ευθύνη. Σα ευχαριστούμε, κυρία Χάιντσλεκ, για τρία λεπτά. Ο συνάδελφο Κούτα, δεν ξέρω μήπω παρέφερε το όνομά σα.